Κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ για να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι δηλώσει Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Επιτροπή σχετικά με τα συμπεράσματα της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης και 29ης Ιουνίου. Καταρχάς θα δώσω το λόγο στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κύριο Ντόναλτ Τούσκ. Καλώς ορίσατε κύριε Τούσκ. Έχετε το λόγο. Thank you. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,